του Συμβουλίου ένα νομοθέτημα σύμφωνα με τη συνήθεια νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού μας ο, ε, ο, ε, τίτλος του νομοθετήματος θα δημοσιευτεί στα πρακτικά της